Πρώτα απ' όλα και πρωτού κάνω τις τελικές μου δηλώσεις θα έλεγα το εξής. Όταν σκέφτομαι το θέμα της καινοτομίας πιστεύω πραγματικά πως πρόκειται για ένα θέμα ε, νοτροπίας και άρα χρειάζεται και κάποια πειθαρχία, να συνεχίζουμε, να μην εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες παρά τις αποτυχίες. Δεν μπορεί να φοβόμαστε την αποτυχία και να θέλουμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τον κόσμο. Φυσικά κάθε φορά που επιχειρούμε κάτι στη ζωή μας, ε, μας διακατέχουν φόβοι. Δεν πρέπει αυτό να μας αποθαρρύνει. Θέλω να φύγετε με αυτήν την εικόνα από εμένα ότι είμαι βαθιά πεπισμένος ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε. Είναι μεγάλη μου τιμή ε, που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Ε, ήμουν βουλευτής, πιστεύω ε, στη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τους βουλευτές και ευχαριστώ και το προσωπικό. που παρακολουθεί την ακρόαση τις τελευταίες ε, τρεις ώρες. Εξίσου σημαντικό, ο μιλητής πολύ ευγενικά ευχαριστεί και εμάς τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ως προς τη μελλοντική μας συνεργασία. Θα είμαι... Θα είναι έντονη η παρουσία μου στο Κοινοβούλιο, διότι μέσα από τη συνεργασία μας μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα. Λέει ένας ε, γνωστός συγγραφέας ε, ότι κανείς από μόνος του δεν είναι τόσο έξυπνος όσο όλοι μαζί. προσπαθήσω κι εγώ να φανώ έξυπνο για να δημιουργηθούν οι ευνοικότερε συνθήκες πλαίσιο. Δεύτερον, για να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης αγοράς εργασίας την έρευνα και να χρησιμοποιηθεί ως θεμέλιο για τις επιστημονικές γνώσεις μας το πάθος, το κίνητρο, η αφοσίωσή μου τόσο στην ιδιωτική όσο και την επαγγελματική μου ζωή σε αυτό το ζήτημα, αλλά κυρίως ο ζήλος και το πάθος που ε, θα ε, προσφέρω ε, κατά την επιτέλεση των καθηκόντων μου, αν με επιλέξετε, θα μου επιτρέψει να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουέβας, οριστής επίτροπος, η έρευνα, επιστήμη και η καινοτομία είναι ύψης της σημασίας για μας. Δημιουργούμε προγράμματα ήδη από τη δεκαετία του 70 και θεωρούμε σε αυτή την Επιτροπή ότι είμαστε υπεύθυνοι για την έρευνα, και καινοτομία αλλά και την εκπαίδευση. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε έναν πρώην φοιτητή Εράσμους ως υποψήφιο, υποψήφιο επίτροπο. Αυτό σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε σε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους της ε, δημόσιας ε, που από δημόσια ε, μέσα μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, τους εκπροσώπους ΜΚΟ, κρατών μελών και ούτω καθεξής. Έχω να σας πω και τα εξής. Αν μπορείτε να παραμείνετε μαζί μας, κύριε Επίτροπε. Ένα καλό νέο. Αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε την ακρόση. 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα λοιπόν. Σήμερα όμως θα συναντηθούν οι συντονιστές στις 3 το απόγευμα και στις 6 επίσης Μετά από δύο ακροάσεις θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Στις 6 το απόγευμα, σήμερα, ε, έχουμε την ακρόαση του κυρίου Σέπκοβιτς. Ε, και όπως ξέρετε συμμετέχουμε και εμείς μαζί με την Επίτροπη Μεταφορών. Έξι λοιπόν μέλη από την Επίτροπή μας θα μεταβούν στην ΤΡΑΝ για να υποβάλουν ερωτήσεις. Αλλά είναι ανοιχτή για όλους και ξέρουμε ότι το, το θέμα των δορυφόρων και των μεταφορών είναι ύψης της σημασίας και για μας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε και τον υποψήφιο επίτροπο. Γεια σας. Great.